Αγαπητοί συνάδελφοι,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 σύμφωνα με τα ισχύοντα περί άμεσης καθολικής εκλογής των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στην έναρξη της πρώτης συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά τις εκλογές. Αγαπητοί συνάδελφοι, να σας παρακαλέσω να σηκωθείτε για τον ύμνο της Ευρώπης. Liebe Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, σας ε, καλωσορίζω εγκάρδια στην ε, πρώτη συνεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά τις ε, εκλογές. Συγχαίρω όσους επανεξελέγησαν και όσους εξελέγησαν για πρώτη φορά. Κάτι λιγότερο από τους μισούς 700, από τους 736 βουλευτές εξελέγησαν για πρώτη φορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ιδιαίτερα ικανοποιητικό είναι το ότι 35% των βουλευτών είναι γυναίκες, το υψηλότερο ποσοστό μέχρι σήμερα. «170 εκατομμύρια πολίτες ψήφισαν στις εκλογές και η δική μας η δουλειά αγαπητοί συνάδελφοι εξυπηρετεί ένα μεγάλο στόχο την ένωση της Υπήρου, της Υπήρου μας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ κατά τη διάρκεια των εργασιών μας πως βασιζόμαστε σε κάποιες αξίες, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ελευθερία, τη δημοκρατία, το δικαίωμα στην ειρήνη. Αυτές είναι οι βάσεις των όσων κάνουμε. Μας συνδέει η αλληλεγγύη θα ήθελα να σας παρακαλέσω αγαπητοί συνάδελφοι πάντα να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Εάν συμβαίνει αυτό θα είμαστε και επιτυχείς. Θα ήθελα να περάσουμε τώρα στο έργο της σημερινής ημέρας. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω πως σύμφωνα με τον κανονισμό υπό την προεδρία του αποχωρούντος Προέδρου δεν μπορεί να γίνει καμία άλλη συζήτηση παρά μόνο η εκλογή του Προέδρου και η εξέταση των εντολών.